Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης, δηλαδή η οθέτηση της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το σχέδιο ημερησίας διάταξης μπορεί να υιοθετηθεί ως έχει. Ανακοινώσεις του Προέδρου. αποστολή στο Ντουβάι τα έγγραφα που συμπεριλαμβάνουν ε, την επίσκεψη στο Ελσίνκι βρίσκονται στα πρακτικά της συνεδρίασης θα υπάρχει διερμηνία σήμερα σε 13 ε, γλώσσες και ως συνήθως μπορείτε τα στοιχεία τα βρείτε για τη συνεδρίαση να τα βρείτε ηλεκτρονικά και θα γίνει και web streaming Θέμα 3. Οι συστάσει του συντονιστή κυκλοφόρησαν ηλεκτρονικά. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης τη 12 η και 13 η Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τα πρακτικά θεωρούνται ως εγκριθέντα. Περνάμε στο 5. Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής για τις διεξαγόμενες διαθεσμικές διαπραγματεύσεις για τις ιατρικές συσκευές και τις διαγνωστικές μεθόδους in Τελευταία συνάντηση έγινε στις 3 Δεκεμβρίου τα αντιθέματα που συζητήθηκαν ήταν δύο διαδικασίες αξιολόγησης. Το Κοινοβούλιο επέβαλε ένα κείμενο συμβιβασμού στο Συμβούλιο, κεφάλαιο 7, σχετικά με την εποπτεία. Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθεί να γεφυρώσει τα δύο άκρα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αυτή διαδικασία και να κρίνεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στο κεφάλαιο 7 παραμένουν εκκρεμοί μόνο ορισμένα θέματα ελάσσονος σημασίας. Το επόμενο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε σε θέματα που εκκρεμούσαν από την προηγούμενη συνάντηση. Η έκτη συνάντηση θα γίνει τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, υπό την Ολλανδική Προεδρία. Ο δεύτερος ε, τρίλογος για τις ε, δραστηριότητες θα αφορά την εφαρμογή στον κλάδο των τροφίμων, ενώ η δεύτερη, που έγινε, ο δεύτερος που έγινε την 1η Δεκεμβρίου έδωσε τη δυνατότητα να συζητηθούν άρθρα και που συμφωνία για ορισμένα βασικά θέματα. Ορισμένα βασικά θέματα που αφορούσαν, αφορούσαν τη συνοχή, αλλά τα θέματα αυτά θέθηκαν για τις επόμενες συναντήσεις. Συζητήθηκαν διάφορες τεχνικές πτυχές του θέματος. Η τρίτη συζήτηση θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου. Ο τέστερος τρίλογος θα αφορά τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα το οποίο συμπεριλαμβάνει αρκετά σημεία που παραμένουν εκκρεμή. Ε, ε, υπήρχε μια μεταβατική περίοδο για τους, ε, ε, τις οποίες υπήρχε συμφωνία από το Συμβούλιο. Επειδή υπήρξε μια αλλαγή άποψης, ε, συμφωνήθηκε να υπάρξει μία νέα πρόταση του Συμβουλίου, μία τεχνική συνάντηση έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου για να συζητηθούν τεκρεμή θέματα συμπεριλαμβάνοντας τις ε, κατεξουσιοδότηση ε, πράξης. Η συνάντηση θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου. Θα μπορούσαμε τώρα να περάσουμε στο θέμα 6 της ημερησίας διάταξης, δηλαδή κανόνας 106, Η ένσταση προέρχεται από διάφορες πολιτικές ομάδες, ΔΙΑΛΤΕ, Πράσινη, ΓΚΟΥΕ, ΕΦΤΗ και θα ήθελα αμέσως να δώσω το λόγο σε αυτούς που ε, έχουν στάσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Απόψε έχουμε να ψηφίσουμε για μια ένσταση πρόκειται για τις real drive emissions, τις ε, πραγματικές εκπομπές ρήπων δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Χρειαζόμαστε αντανάκλαση των πραγματικών συνθήκων οδήγησης καλύτερα στο δρόμο για αυτές τις μετρήσεις. Ελαστικότητες που έχουν οι σημερινές δοκιμασίες δεν πρέπει να υπάρχουν ελαστικά περιθώρια. Έχουμε το Ευρω 5 και Ευρω 6 και ήμουν ο ίδιος εισηγητής για το 2007-2008 για αυτή την υπόθεση Δηλαδή έχουμε νομοθεσία που προωθήσαμε τελικά, όπου όλα αυτά τα θέματα αγωνιστήκαμε να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για να τα προαγάγουμε. Αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό εγκρίθηκε η νομοθεσία. Σε πρώτη ανάγνωση Ευρω 5, 180 για τα νόξ, οξύδια του αζότου και στη συνέχεια Ευρω 6, πράγμα το οποίο άρχισε να ισχύει φέτος ως νέο ε, πλαίσιο Ευρω 6. Στόχος μας ήταν να τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές βέβαια. Σίγουρα οφείλεται στο ότι πόσο ένας ή άλλος οδηγός παταγκάζει και έτσι χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ταχύτητα και έτσι έχουμε μεγαλύτερες εκπομπές ρήπων ενδεχόμενα. Ακούσαμε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέβαλε 1,6 ως αξία, ως συντελεστή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εμείς ρωτήσαμε πώς συντίθεται αυτό ο συντελεστής. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφήνεια μας είπαν επιστημονικά τεκμηριώνονται όλα με αυτόν τον τρόπο και έχουν υπολογιστεί όλα και έτσι με τους νέους υπολογισμούς αυτός πρέπει να είναι ο συντελεστής. Και η Τεχνική Επιτροπή αποφάσισε ότι έχουμε ένα συντελεστή επιδίνωσης 2,1. Δηλαδή υπέρβαση κατά 210% του περιθωρίου εδώ δεν πρόκειται μόνο για το θέμα της νομοθεσίας. Επ' αυτού μπορεί να έχει κανείς διαφορετική άποψη. Ο ένας μπορεί να θέλει το Ευρω 5, ο άλλος μπορεί να προτιμά το Ευρω 6 ως πλαίσιο. Πρέπει όμως να προσέξουμε αυτά τα οποία εγκρίναμε και αποφασίσαμε κάποτε, τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο να ανταποκρίνονται λειτουργικά σε αυτά τα οποία νομικά και νομοθετικά προβλέπονται και πρέπει να εφαρμόζονται. Και 210% υπέρβαση ενός συντελεστή που εμείς εγκρίναμε. Ε, πώς θα το εξηγήσω αυτό σε έναν πολίτη. Και πρέπει να είμαστε εκ του σύνεγγυς πάρα πολύ κοντά στα πράγματα. Γι' αυτό η ομάδα μας μετά από έντονες διαβουλεύσεις είπε αυτός ο συντελεστής 2,1 δεν μπορεί να γίνει δεκτός έτσι ως έχει. Και μακροπρόθεσμα ότι δηλαδή δεν θα είναι χρονικά περιορισμένο αυτό, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε ούτε αυτό. Αν έχει επιτυχία η ένσταση απόψε, θα μπορέσουμε στο μεσοδιάστημα ίσως ε, να καταφέρουμε να μπορέσει να υπάρξει διαπραγμάτευση επιπρόσθετη ώστε να μην γίνει αυτό πραγματικότητα τελικά. Χρειαζόμαστε πραγματικών συνθήκων δοκιμασίες, υπό πραγματικούς όρους δοκιμασιών. Το χρωστάμε στους πολίτες μας αυτό και γι' αυτό εμείς ως ομάδα υποστηρίζουμε την ένσταση απόψε. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκεμπράντη παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Ευχαριστώ πρόεδρε. Συζητήσαμε αυτό το θέμα στο παρελθόν. Δεν χρειάζομαι πολύ χρόνο λοιπόν γι' αυτό. Κάποιες παρατηρήσεις ε, σε θέματα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη. Σε μια χρονική στιγμή όπου τα αυτοκίνητα προκαλούν την κυριότερη ρήπανση της ατμοσφαίρας ε, και όταν δεν συνάδουν και δεν ευθυγραμμίζονται με τα πραγματικά νομικά όρια που πρέπει να ισχύουν έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη στις πόλεις μας ώστε να διασφαλίζουμε καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα στις πόλεις μας για τους πολίτες μας. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα λοιπόν σε αυτό το πεδίο. Δεύτερον, για τους φιλελεύθερους αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να υποβάλουμε ένσταση. Θέλουμε δίκαιο ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί αυτοκίνητοι το βιομήχανη που συμμορφώνονται με τους κανόνες και κανονισμούς των νομοθετών. Με το να αναβάλουμε λοιπόν έτσι την επιβολή αυτών των ορίων, επιτρέποντας περιθώρια σε εκείνες τις εταιρείες που ιδιαίτερα εξαπατούσαν και εξαπάτησαν και να αφήσουμε χρόνια ώστε το 2,1 να ισχύει 210% δηλαδή υπέρβαση ε, δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιο ανταγωνισμό με τέτοια κατάσταση και τέλος πρόεδρε είναι επίσης ένα ζήτημα των σωστών δημοκρατικών διαδικασιών που πρέπει να ισχύουν. Οι σωστές δίκαιες δημοκρατικές διαδικασίες και διεργασίες πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και κανονισμούς. Δεν νομίζω ότι είναι τεχνικού χαρακτήρα απόφαση που μπορεί να λαμβάνεται από μια τεχνική επιτροπή. Είναι υψηλότατος ο βαθμός πολιτικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η δημοκρατία μας να, λειτουργεί με τέτοιες ελλείψεις. Δεύτερο, για τη δημοκρατική διαδικασία, η απόλυτη απουσία διαφάνειας τα κράτη-μέλη δεν ήταν διαφανή στις θέσεις που, που υιοθέτησαν στις 28 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες τέλος τέλος έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουν οι κυβερνήσεις τους, πώς τοποθετούνται και για ποιο λόγο στις Βρυξέλλες. Δεν είναι όμως διατεθειμένες οι κυβερνήσεις να διασφαλίσουν διαφάνεια. Δεν υπάρχει καμιά δικαίωση και δικαιολογία για μια τέτοια απόφαση και δεν υπάρχει καθόλου οποιαδήποτε λογοδοσία, δημόσια λογοδοσία στη συνέχεια υστερότερα από πλευρά των κρατών μελών. Αυτή είναι η κυριότερη λόγη για του φιλελεύθερου, που καταθέσαμε την ένσταση και υπερψηφίζουμε την ένσταση. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now for GUE, e, Ευχαριστώ για την ενωτική αριστερά, η κυρία Κιλόνεν, παρακαλώ. Hyvät kollegat, GUE-NGL-ryhmä Μικροφωνίζει και δεν ακούγεται. Εμεί Εμείς στηρίζουμε αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Δεν ακούγεται η διερμηνία επειδή μικροφωνίζει. Πρέπει να σας πω πως ε, το όργανο αυτό ε, με συγχωρείτε, διακόπτει η ομιλήτρια, υπάρχει πρόβλημα με την αγγλική μετάφραση. Έτσι κι αλλιώς πάντα όλοι προβλήματα έχουμε. Okay. Do you want me speak Finnish or English or? Να μιλήσω φιλανδικά, αγγλικά. You can start another time. English works. now. Yes. Okay. okay. Yeah. yeah, I, I can finish already. yeah. yeah. Hyvät puheenjohtaja, hyvät kollegat. Marista. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ε, tota λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τροποποίησει σε ένα κανονισμό οι οποίες αντίκενται και στο γράμμα και στο πνεύμα του σημερινού κανονισμού. Δυστυχώς με τον τρόπο αυτό ξεπερνάμε ε, ακόμα και το περιθώριο λιγμών που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις με τους συντελεστές που έχουμε στον κανονισμό και αν επιτρέψουμε να υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ πραγματικών συνθήκων και εργασιακών συνθήκων και σε πέντε χρόνια από το 2,1 προσθέσουμε ακόμα 0,5% τότε θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση η οποία δεν θα σέβεται τους τρέχοντες περιορισμούς στις εκπομπές και θα ήθελα να πείτε και στην περίπτωση αυτή πότε θα καταλήξουμε σε τιμές οι οποίες σε τεχνικό επίπεδο θα είναι εφικτές. Αυτό το οποίο απαιτούμε εμείς είναι μία καινούργια πρόταση κανονισμού που θα τη βάλετε στο τραπέζι μπροστά μας και όπου η λήψη απόφαση θα γίνει με δημοκρατικό τρόπο, γιατί μιλάμε για ανθρώπινη υγεία, μιλάμε για περιβάλλον και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει ε, να προστατευτούν στο μέγιστο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά έχουν ήδη υποθεί. Θα ήθελα απλώς να τονίσω Αυτό που θέλω να τονίσω λοιπόν είναι πως ο σκοπός μας εδώ, σε νομοθετικό επίπεδο, είναι να έχουμε ε, πιο αυστηρά όρια εκπομπών και για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν βενζίνη και για αυτά τα οποία χρησιμοποιούν δίζελ. Είπα 0,8 για κάθε χιλιόμετρο. Όσοι νομοθέτες θέσαμε αυτό σε στόχο. Πριν από πολλά χρόνια η ίδια απόφαση όταν ε, αποφασίσαμε το Euro 6 είναι πως έχουν 6 χρόνια για να εφαρμόσουν αυτές τις τιμές και παράλληλα αποφασίστηκε πως θα πρέπει να κάνουμε δοκιμές για τις πραγματικές εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες. Ήδη τότε ξέραμε από τότε πως νέες δοκιμές θα αναπτυχθούν και μπορεί να γίνει μια τεράστια συζήτηση για ποιο λόγο χρειάζεται τόσο χρόνο να ετοιμάσει αυτές τις νέες δοκιμές η Κομισιόν. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, είναι πια διαθέσιμες και το 2014 τα οχήματα θα έπρεπε, τουλάχιστον τα καινούρια, να συμμορφούνται με τα 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο. Το είχαμε αποφασίσει αποφασίσει εμείς στα πλαίσια της δράσης μας ως συνομοθέτη. 1η Δεκεμβρίου λοιπόν πέρσι 1η Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, πέρσι, θα έπρεπε όλα τα νέα αυτοκίνητα στην αγορά να σέβονται το 0,80 ε, μιλιγκράμμ τα χιλιόμετρα. Στη ΣΥΠΑ αυτά τα πρότυπα είναι στα 40 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο και στην Καλιφόρνια είναι 35 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο. Και ξέρετε πως η αυτοκινητοβιομηχανία σε κάποιο βαθμό καταφέρνει και συμμορφώνεται με τι απαιτήσει των Αμερικανών στη ΣΥΠΑ. Αυτό λοιπόν ο κατασκευαστικό κλάδο τη αυτοκινητοβιομηχανία που προσπαθεί να πείσει εμά πω είναι αδύνατο να σεβαστούν αυτού του περιορισμού, θα έπρεπε να μα εξηγήσουν για ποιο λόγο μπορούν στη ΣΥΠΑ και με τα οχήματα diesel. Ξέρουμε πως έχουν λιγότερα από εμά, αλλά τα οχήματα diesel που κυκλοφορούν στη ΣΥΠΑ κυκλοφορούν με αυτό τον περιορισμό εκπομπών, άρα γίνεται. Και είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι που προσπαθούν να μας πιέσουν να ανεβάσουν τα όρια και τις τιμές στην Ευρώπη και όχι οι τεχνικοί λόγοι που τους υποχρεώνουν ε, στο να μας ζητούν κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει τώρα. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν να χαλαρώσουν τα επίπεδα μέσω μιας τεχνικής επιτροπής η οποία χρησιμοποιεί ένου είδους συντελεστή συμμόρφωσης. Εδώ όμως έχουμε δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα. Καταρχήν, γιατί χρειάζεται μεταβατική περίοδος, γιατί τα νέα αυτά όρια θα είναι ε, ενισχύ από το 2021 και μόνο και η εφαρμογή θα επεκταθεί ε, μέσω μιας τεχνικής επιτροπής, ενώ τότε πριν από χρόνια αποφασίσαμε πως δεν χρειάζεται και πως θα συμμορφωθούμε το 2014. Και δεύτερον, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ο συντελεστής συμμόρφωσης μετά από το 2021 να είναι στο 1,5%. Δηλαδή κάθε όχημα δίζελ θα επιτρέπεται να εκπέμπει 120 μιλιγκράμμ το χιλιόμετρο. Και στην Τεχνική Επιτροπή το μόνο που κάνουν είναι να νερώνουν ένα όριο το οποίο αποφάσισαν οι συνομοθέτες πριν από πολλά χρόνια. Εμείς ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπέβαλε πρόταση να μας εξηγήσει για το γεγονός ότι χρειάζεται αυτή η παράταση της ε, περίοδου εφαρμογής και γιατί ζητούν υψηλότερες τιμέ Και μας είπανε ναι γιατί χρειαζόμαστε περιθώριο στατιστικού λάθους λόγω των νέων δοκιμών. Μα στην πρότασή τους μας είπαν και τα επιχειρήματά τους είναι πως το στατιστικό περιθώριο θα πρέπει να είναι 1,18. Αυτός δεν είναι ο συντελεστής που επιτρέπουν και τα κράτη-μέλη σε πολιτικό επίπεδο αποφάσισαν 1,5. Είναι πολιτική απόφαση και ελήφθη μέσω μιας τεχνικής επιτροπής. Οπότε ακόμα και αν σε πολιτικό επίπεδο εσείς συμφωνείτε με κάτι τέτοιο που θα ήταν περίεργο γιατί πριν από χρόνια δεν το δεχόσασταν σε πολιτικό επίπεδο αλλά ακόμα και αν τώρα πολιτικά συμφωνείτε με τα όρια αυτά δεν μπορείτε να επιτρέψετε μια τέτοια απόφαση να λαμβάνετε σε τεχνική επιτροπή χωρί να υπάρχει ρόλο για εμά το Κοινοβούλιο ω συνομοθέτη. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παρακαμφθεί και νερώνεται ένα πρότυπο σε μια τεχνική επιτροπή. Νομίζω αυτή είναι αρκετή λόγια έτσι ώστε να έχουμε αντιρρήσει για το συγκεκριμένο. Και φαντάζομαι πως και όλες οι πολιτικές ομάδες εδώ στην αίθουσα σε πολιτικό ρόλο θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα αντιτεθούν σε ε, αυτού του είδους τη χαλάρωση των κανόνων και της ε, μη εμπλοκής του συνομοθέτη γιατί αυτό διακυβεύεται εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ παρά να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπαν οι συνάδελφοι μέχρι τώρα. Η Ιταλική Αντιπροσωπεία της ομάδας FTD υποστηρίζει αυτή την ένσταση. Νομίζω ότι οι λόγοι παρατέθηκαν εκτενώς από τους συναδέλφους. Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που ήδη υπόθηκε, ότι πρόκειται για μια σημαντική τροποποίηση μιας βασικής νομοθετικής πράξης και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, γιατί υπάρχουν τεχνικές επιτροπές πρότειναν και προωθήθηκαν θέσεις που είναι αμυγός πολιτικές, συνεπώς σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να παραμείνει η συζήτηση. Εξάλλου με, τα καινούργια, με τις καινούργιες αυτές δοκιμές το μόνο που κάνουμε είναι το να κάνουμε περισσότερες παραχωρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες και μολύνουν αλλά και εξαπάτησαν δύο φορές τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό όλες οι πολιτικές ομάδες να συμφωνήσουν με αυτή την έσταση που θα ψηφιστεί σε λίγο. Ευχαριστώ. Κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμένα η άποψή μου είναι διαφορετική. Ξέρετε ότι η ομάδα μου δεν έχει προσυπογράψει αυτό το κείμενο. Δεν αφορά μια διαφορετική άποψη ως προς την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Δεν είναι διαφορετική άποψη γιατί θέλουμε να, γίνει κάτι με τις, δοκιμασ... με τις δοκιμές αυτές. Συμφωνώ με αυτό. Θέλω να πω στα μέλη τι κάνουν όταν απορρίπτουν αυτό το κείμενο. Είναι ένα θέμα πολιτικό, βεβαίως. Αλλά θα πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι κάνουμε. Θα καθυστερήσουμε την εισαγωγή του ΑΤΗ. Γιατί αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή η συμφωνία τον Οκτώβριο είναι η συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου ότι δέχονται να περάσουν από την άλλη συμφωνία στο αντί σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα καινούριο ε, τύπος δοκιμών. Βεβαίως συμφωνήσαμε ότι η βασική αρχή βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη Συμφωνία Τεχνικής Επιτροπής που αφορά το αντί της πραγματικές εκπομπές ε, ρήπων. Ελπίζω λοιπόν αυτά τα σημεία να τονιστούν το συντομότερο δυνατό και νομίζω θα, δούμε, πρέπει να δούμε πώς φτάσαμε στους, στα σημεία συμμόρφωσης. Είναι απόλυτα δυνατόν το να μην προβάλλει αντιρρήσεις γι' αυτό, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εμεί η Επιτροπή σε συνδυασμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή γιατί από πλευράς Συμβουλίου υπάρχει επιθυμία διαπραγμάτευσης είδαμε τι είχε τεθεί επιτάπητο, δηλαδή υπήρχε διάθεση να υπάρξει συναπόφαση από πλευράς του Κοινοβουλίου αυτό το απορρίψαμε εγώ δεν ήμουν παρούσα αλλά από ό,τι κατάλαβα περίφθη από το Κοινοβούλιο Υπάρχει όμως η βούληση και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχει τρόπος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη συμφωνία. Δηλαδή να περάσουμε τώρα στο το αντί στις πραγματικές εκπομπές ρήπων. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει και μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε κάτι την 1η Απριλίου, μέχρι την 1η Απριλίου. Μπορούμε να το ζητήσουμε, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να μας το δώσουν. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μία καθυστέρηση, Έξι μήνες, 12 μήνες. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Τώρα, Ενδεχομένως η απόρριψη, η ένσταση θα μπορέσει να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, αλλά δεν μας βοηθήσει να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Κοιτάξτε την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής. Αν δείτε το άρθρο το εκτιμώντα 14, η Επιτροπή θα εξετάζει τα προβλεπόμενα από το RDE και θα τα ε, προσαρμόσει τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές. Κατά τον ίδιο τρόπο η Επιτροπή θα ελέγχει το επίπεδο συμμόρφωσης και θα καταγράφει τεχνική πρόοδο. Θα εξετάσει τις δύο εναλλακτικέ μεθόδους ε, αξιολόγησης των δεδομένων PM. Αυτά είναι τα ε, ε, στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό το θέμα της συμμόρφωσης. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό, θα πρέπει να μιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα, για το πού θα οδηγηθούμε με τη συναπόφαση και είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό που πιστεύω είναι ότι τα απορρίπτοντας αυτά και λέγοντα ότι δεν το θέλουμε πάλι πίσω, δεν θα έρθει πίσω για μήνες ολόκληρε. Αν θέλετε να κάνουν κάτι οι αυτοκινητοβιομηχανίε, αυτό είναι, ε, ε, αυτό είναι ακριβώς αυτό που δεν θα πρέπει να κάνουμε, γιατί θα περνάει ο καιρός και δεν θα γίνεται τίποτα. Θα ζητούσα λοιπόν από τα μέλη ιδιαίτερα προσεκτικά. Νομίζω ότι λαμβαντής υπόψη ότι υπάρχει στήριξη, θα πρέπει εμείς ως πολιτική ομάδα να θεωρήσουμε ότι είναι επιτακτικό το να δώσουμε μία εναλλακτική λύση και να μπορούμε να έχουμε άποψη για τον παράγοντα της συμμόρφωσης. Now... Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ είχαμε του ήπιου λογισμικού το σκάνδαλο και αυτό φυσικά ανησύχησε και είναι απόλυτα δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο και ότι δεν θα δημιουργηθούν μειονεκτήματα για την Ευρώπη ως έντρα βιομηχανιών. Αυτό που πρέπει λοιπόν να πράξουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι οι νέες διεργασίες που θα αρχίσουν να ισχύουν θα, ισχύουν, θα αρχίσουν να ισχύουν το 2016 και όχι από το 2017 όπως αναφέρθηκε. Από πλευρά στον ΗΠΑ τώρα υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές και αυτό αφορά και τα, τις πλωτές μεταφορές και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται εκεί. Κατηγορούμαστε ότι εμείς ε, ότι έχουμε εκπομπές τρύπων ε, ιδιαίτερα ρηπαντικές, ε, μολύνουσες. Όμως όταν έχουμε υπέρβαση κάποιων τιμών πρέπει να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός ουσιώδη τμήματα του κανονισμού από πλευράς του 2007 80 μιλιγκράμμα όσον αφορά την κάλυψη χιλιομετρικών αποστάσεων είναι αυτό περί του οποίου πρόκειται 110% υπέρβαση όμως και μετά το 2020 χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη κάτι τέτοιο να τεκμηριώνεται και να δικαιολογείται επιστημονικά είναι εντελώς εσφαλμένη λοιπόν αυτή η διαδικασία και αυτή η απόφαση να συνεχίσουμε έτσι Μπορεί να υπάρχει κάποια διακύμανση 25%. 25% ε, είναι υπερβολικά υψηλή διακύμανση καταλήτες μπορούν να ενταχθούν ε, με ένα πρόσθετο κόστος που μπορούν να ενταχθούν στον εξοπλισμό ενός αυτοκινήτου και θα δίνει τη δυνατότητα ο καταλήτης να σέβονται αυτές τις τιμές ε, για τη μείωση των ε, ρηπαντών και των εκπομπών. Πρόκειται λοιπόν για χρήματα και δαπάνες που ρυθμίζουν τα πάντα, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες που θα έπρεπε να πριτανεύουν. Οι εκπομπές ρήπων λοιπόν που έχουν ε, ε, ε, επιπτώσεις και στη βιομηχανία δεν πρέπει να, να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και σταθμά γιατί και στη γεωργία θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την κατάσταση όσο έχει σήμερα. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτή η περιβαλλοντική συμφωνία των Παρισίων θα υπονομεύεται με αυτόν τον τρόπο. Αρνούμε να το δεχτώ αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα και οι αποπράσεις συντονιστού υπήρχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις και η σημερινή απόψινή συζήτηση καταδεικνύει πόση μεγάλη ανάγκη υπάρχει να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα από πλευρά μας. Υπάρχουν επιχειρήματα που αποβαίνουν υπέρ, τέλος, ε, ε, καταβαίνουν υπέρ ε, υπέρ της τοποθέτησης ίσως της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς από πλευράς του θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να εξεταστούν αυτά τα πράγματα δεδομένης της γενικότερης πολιτικής συζήτησης μια και περισσότερα ερωτήματα αναφύονται από τις απαντήσεις που δόθηκαν και δεν επαρκούν. Χρησιμοποιήθηκε και το επιχείρημα των αυξημένων τιμών ε, ρήπαντων που οικονομικά λέει οφείλεται σε οικονομικά επιχειρήματα. Εφόσον στην Ευρώπη Ευρώπη ένα οικονομικό και κοινωνικό σύστημα υψηλής ποιότητας διασφαλίζεται πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται με αυτές τις τιμές. Προέρχονται λοιπόν από τη βιομηχανία και αυτό είναι ένας λόγος που πρέπει να μας κάνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη βιομηχανία και τους βιομηχανικούς κύκλους. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, σύνετοι και δίκαιοι. Σημαντικό είναι ο στόχος να τηρηθεί για την μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Εμείς από πλευράς του ΕΛΚ χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για αυτή τη συζήτηση. Δεν θα υποστηρίξουμε ενεργά λοιπόν αυτή την ένσταση. Πρέπει να προετοιμαστούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πλειοψηφικά θα απόσχουμε αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη στην Ολομέλεια και για τον επόμενο καιρό και την επόμενη εβδομάδα να υπάρξουν συζητήσεις που θα διεξαχθούν. Ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση, ότι πρόκειται δηλαδή για μια καθυστέρηση περισσότερο για την βιομηχανία και την οικονομία που χρειάζονται νομική ασφάλεια, νομική βεβαιότητα και οι μεγάλες χρονοβόρες διαδικασίες πρέπει να, να κλείσουν πια. Αν η ένσταση θα είναι το σωστότερο μέσο, αυτό ε, πρέπει να απαντηθεί και απομένει προς απάντηση. Εμείς θα απόσχουμε. Αναμένουμε συζήτηση, περισσότερη συζήτηση από αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι σε μια εξαιρετικά ιδιάζουσα κατάσταση γιατί έχουμε αφενός την καλή θέληση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να μειώσει το βάρος στην αυτοκινητοβιομηχανία γιατί αυτές οι απαιτήσει δημιουργούν ένα υπερβολικό και πολύ αυστηρό σύστημα και ανοίγουν την πόρτα σε προσπάθειες να παρακαμφθεί η νομοθεσία. Όμως η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σέβεται τη δημοκρατική διαδικασία, την κοινοβουλευτική διαδικασία. Έχω ήδη εκφράσει την άποψή μου. Θα πρέπει να θυμάται η Κομισιόν πως τα συμφέροντα των κρατών μελών και των οικονομιών τους θα πρέπει να είναι ε, πιο σημαντικά από τις φρενήρες προσπάθειες νομοθεσίας σε όλους τους τομείς. Εμείς θα είχαμε συμφωνήσει με την Κομισιόν αν είχε σεβαστεί τη διαφάνεια και τη δημοκρατική διαδικασία. Γι' αυτό η δική μας ομάδα δεν θα συμμετέσχει, δηλώνουμε αποχή από αυτή την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, δεν βλέπω άλλους να ζητάνε το λόγο. Η κυρία Κατρίνη, παρακαλώ. Πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όσα είπε η συνάδελφος Γκέρλινγκ γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν εμείς ψηφίσουμε κατά για λόγους συναισθηματικούς ή με έναν παρορμητικό τρόπο, στην ουσία θα αναβληθεί η υιοθέτηση μέτρων που δίχως άλλο θα είναι χρήσιμα για την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας άκουσα μερικά πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ απόλυτα γιατί όταν κάνουμε μια σύγκριση με τις εκπομπές στην Αμερική είναι λάθος. Εκείνοι αναφέρονται στα μέσα όρια, εμείς στα μέγιστα όρια. Το να συγκρίνουμε το μέσο με το μέγιστο των εκπομπών έχω την εντύπωση ότι δεν είναι σωστό. Μου λέτε όχι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω και θα πρέπει να πω ότι ενημερώθηκα αρκετά πριν το πω. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε συγκρίσεις. Είναι αλήθεια ότι όλοι μας έχουμε στόχο την ποιότητα του αέρα και την υγεία των συμπολιτών μας. Κατά την άποψή μου, επειδή θα πρέπει να συζητήσουμε και να βελτιώσουμε τα πάντα, το να απορρίψουμε, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι προθέσεις ε, δεν με αρκούν, ε, θα επιτύχουμε ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω αν ε, τελικά θα απόσχω, ενδεχομένως θα καταψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ, Σε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θεωρώ σε μερικά από τα σημεία που άκουσα. Η Επιτροπή μας έδωσε ορισμένα δεδομένα. Μήπως θα μπορούσε κανείς να μας πει για ποιο λόγο θα πρέπει να δεχτούμε τα υψηλότερα όρια που θέτει η Επιτροπή και θα πρέπει να δεχτούμε ότι το αποτέλεσμα της απόφασης είναι κακό, τα όρια αυξήθηκαν, εδώ ακούσαμε για μέσες ή για υψηλές και υψηλότερες τιμές. Επίσης γνωρίζουμε ότι η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία μεταθέτει το ρόλο του Κοινοβουλίου και γίνεται ένας συμβουλευτικός φορέας και όχι ένας φορέας που συναποφασίζει. Η απόφαση έγινε την, ε, λήφθη μέρα που γινόταν μια γενική απόφαση και ζητήθηκε από όλες τις ομάδες να πάρουν θέση. Η απόφαση υιοθετήθηκε στις Βρυξέλλες. Καταλαβαίνω ότι είπε η Τζούντι Γκάρλεν σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη καθυστέρηση. Πιστεύω ότι τώρα η κατάσταση διαφέρει σε σχέση με το 2007. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που ε, αφορά ε, τις πίσω σελίδες εξειδικευμένων δημοσιευμάτων. Αυτό είναι ένα καθημερινό θέμα, ένα θέμα που βρίσκεται, γίνεται πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες. Ε, Σήμερα υπάρχει ένα άρθρο στην Guardian. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν το θέμα, καταλαβαίνουν τις επιπτώσεις που θα έχει και οι ίδιοι οι αυτοκινητοβιομηχανοί θα αρνηθούν να, ε, συνεργαστούν. Αλλά αυτό δεν δείχνει σωστά το ρόλο που έχει το Κοινοβούλιο στην επίλυση αυτού του ε, θέματος. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ αυτής της ένστασης. Ευρωπαϊκή Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Πολύ προσεκτικά ακούσαμε όλες τις ανησυχίες που εκφράστηκαν απόψε και τις παίρνουμε όλες με πολύ σοβαρά. Απόλυτα σεβόμαστε οποιαδήποτε απόφαση ίσως ε, μπορούσε να ληφθεί σήμερα. Όμως επιτρέψτε μου να επεξηγήσω την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την νομοθεσία αυτή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι απόλυτα συμμεριζόμαστε τον ίδιο στόχο και εμείς. Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξίσου και εμείς θέλουμε να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο, ώστε να συμμορφώνονται οι κινητήρες και τα αυτοκίνητα diesel με μηχανές εσωτερικής καύσης για τα οξύδια του αζότου ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται. Αυτός είναι ο κοινό στόχος που όλοι έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα πώς θα επιτευχθεί αυτός ο κοινό στόχος. Εμείς θεωρούμε σε Επιτροπή ότι η απόφαση που ελήφθη από την Τεχνική Επιτροπή στις 28 Οκτωβρίου μας φέρνει πιο κοντά στο να πετύχουμε τη μείωση των ε, οξυδίων του αζότου νοξ Ακούμε ότι υπάρχουν υπερβάσεις 50%, 20% αληθεύει αυτό. Όμως αυτή η απόφαση σε σχέση με την, τον συντελεστή 2 δεν πρέπει να το ξεχνάμε τι συμβαίνει με τα οξύδια του αζότου. Και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του πλαισίου Ευρω 6 και αν δεν γίνεται αυτό θα πρέπει να υπάρξει ε, δράση που θα, αναλάβει, θα αναλυφθεί. Θεσπίζοντας αυτά θα πρέπει να υπάρξουν και πρόσθετες δοκιμές, πειραματικές δοκιμές. Αυτό αποτελεί τμήμα αυτού του πλαισίου και αυτό είναι ο λόγος σήμερα για να διασφαλίσουμε ότι όρια εκπομπών που καθορίζονται από το Ευρω μας οδηγούν στο να μεταθέσουμε από τα πειραματικά, τις πειραματικές δοκιμές στις πραγματικές δοκιμές με όρους πραγματικής λειτουργίας αυτές τις δοκιμασίες. Υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό του νομικού συστήματος που υφίσταται και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής που ελήφθη πριν από δύο μήνες καθορίζει αυστηρά περιθώρια που με κανένα τρόπο δεν αλλάζουν, δεν αλλοιώνουν ή δεν υπερβαίνουν τα ρυθμιστικά πλαίσια του Ευρω 6. Συμπληρώνουν ή παραπληρώνουν αυτό το πλαίσιο και για πρώτη φορά αυτό είναι ουσιώδης διαφορά σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Είναι η πρώτη φορά οποτεδήποτε για την εισαγωγή αυτού του συστήματος ε, δοκιμασιών εκπομπών ρήπων με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι με τις πραγματικές ε, συνθήκες λειτουργίας αυτό είναι ένας συντελεστής που κάνει, αναγκάζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κινηθούν ακόμα περαιτέρω. Αν υπήρχαν αυτές οι, αυτοί οι κανόνες δύο ή τρία χρόνια αργότερα, η πρόοδος που επιτυγχάνεται σήμερα δεν θα είχε επιτευχθεί. Αυτό είναι σαφές συμπέρασμα για το τι θα συνέβαινε με οποιαδήποτε καθυστέρηση για περαιτέρω αλλαγές. Τώρα, ότι χρειάζεται συμβιβασμό που αναφέρατε, ορθό αυτό, αλλά η απόφαση δεν λαμβάνεται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητείται το θέμα με τα κράτη-μέλη και λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη-μέλη τα θέματα αυτά στι απόψει του. Ακόμα και αν υπάρχει ένα συμβιβασμό, ο συμβασμός αυτός εντάσσεται στα εφικτά όρια που αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ακριβώς της λύσης κάνοντας λόγο για αυτά τα ζητήματα όπως επαρκώς επεξηγήσαμε αξιολογήσαμε με τις υπηρεσίες μας τα θέματα αυτά και είπαμε ότι η αύξηση στο 2,2 μπορεί να οδηγήσει παρόλα αυτά στο να επιτευχθούν οι στόχοι που είναι ευκταίοι. Αποτελεί ένα συμβιβασμό λοιπόν. Μόλις ξεκινήσαμε με πολύ, ξεκινήσαμε με πολύ πιο φιλόδοξες ε, ε, προοπτικές ε, και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι λόγοι για τους οποίους υπήρξαν και τα ερωτήματα. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε να υπάρξει αυτή η περίοδος προσαρμογής και λόγω των στατιστικών ισοσφαλμάτων ή παρατυπιών. Κάνουμε λόγο για μια απόλυτα νέα και νοφανή τεχνολογία. Είναι η γραμμή αφετηρίας αυτή. Δεν είναι η γραμμή τέρματος. Δεν τερματίζουμε με αυτό το σημείο. Ξεκινάμε μόνο και γι' αυτό θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο με τις προτάσεις μας ε, στη δέσμη μέτρων τοποθετηθήκαμε έτσι. Να λάβετε υπόψη ότι αυτή η ρήτρα αναθεώρησης ε, σημαίνει ότι καμιά αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα προετοιμάσει ή δεν θα εισαγάγει τεχνολογία που θα πρέπει να είναι εξορισμού περιορισμένης διάρκειας, προσωρινή Γι' αυτό οι αυτοκινητοβιομηχανίες προετοιμάζουν τεχνολογίες και προοπτικές που μελλοντικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγήσουν θα ευθυγραμμιστούν με αυτές τις ε, ε, διατάξεις. Το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή πρέπει να μας κάνει να πούμε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει μέσα σε περίοδο 2-3 ετών να μειώσουν τους ρήπους τους. Υπάρχει λοιπόν πολύ σημαντικό κίνητρο να μπορέσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες πέρα από το 1,1 να μπορέσουν να προχωρήσουν. Είναι απόλυτα πεισμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να παραμείνουμε στους ε, όρους αρμοδιοτήτων μας ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις δοκιμασίες αυτές ε, όχι, σε πειραματικά, ε, όχι πειραματικά αλλά σε ε, υπόρους πραγματικής λειτουργίας. Και θα πρέπει να πούμε, μπορεί αυτό να μην είναι το τελικό ευκταίο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει. Και η ένσταση ζητεί να υπάρξουν νέες δοκιμασίες από την Κύπτροπη το πρώτο ερώτημα εδώ. Πραγματικά σε ποιο μέτρο και βαθμό θα είμαστε ικανοί να το πράξουμε αυτό. Αυτά όλα πρέπει να συζητηθούν φυσικά με τα κράτη-μέλη. Πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη σε δεύτερο γύρο επ' αυτών των θεμάτων. Να δούμε τι θα γίνει με τις φιλοδοξίες που έχουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγηθούμε σε καλύτερα αποτελέσματα, σε αποτελέσματα που θα ικανοποιήσουν όλους όσους έχουν κάποιες αμφιβολίες και υπάρχει και μια δεύτερη εναλλακτική λύση, συναπόφαση. Αν κάνουμε λόγο για την δυνατότητα για τη διαδικασία συναπόφασης δεν θα κάνουμε λόγο για καθυστέρηση έξι μηνών αλλά για καθυστέρηση δύο ή τριών ετών και υπάρχουν πράγματι εδώ προβλήματα σε σχέση με αυτή την καθυστέρηση. Να προβληματιστούμε να δούμε πού θα οδηγηθεί η κατάσταση με αυτή την ένσταση τελικά και ποια τροπή θα πάρει. Και κάνοντας λόγο τώρα για την δέσμη μέτρων, ευρωδέσμη μέτρων, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που εξετάζουμε, αντιμετωπίζουμε τα θέματα των οριακών τιμών, των όρων συμμόρφωσης ε, και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το εξειδικευμένο τμήμα της νομοθεσίας, δεν πρέπει να στερηθούμε δύο πολύ σημαντικά εργαλεία το ένα το οποίο αφορά τις ε, συσκευές ε, και τον εξοπλισμό, διότι πραγματικά η δική μας νομοθεσία είναι οι μόνοι κανόνες και κανονισμοί που θα ε, δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και εισάγεται σε σχέση με ένα σύστημα το οποίο υφίσταται στη ΣΥΠΑ και που έχει συζητηθεί. Δηλαδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να δηλώνουν ποιες είναι οι στρατηγικές τους για τις εκπομπές ρήπων. Αυτό δεν αποτελεί τμήμα αυτού του πλαισίου για μας σήμερα. Και έτσι αυτό εν μέρει ίσως μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση με την Volkswagen. Δεν κάνουμε λόγο μόνο για δοκιμασίες ε, και τιμές, αλλά για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο σε σχέση με το αν δεν προχωρήσουμε έτσι θα μας οδηγήσει στο να στερηθούμε από αυτά τα μέσα ενδεχόμενα. Αυτά είχα να πω από πλευρά τη Επιτροπή σε αυτή τη φάση. Και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε μετά τη συζήτηση στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης για, την, ε, για το ψήφισμα αυτό και την ψηφοφορία του. Έχουμε λάβει λοιπόν ένα αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Χρειαζόμαστε 19 μέλη να εκφραστούν υπέρ της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ποιος στηρίζει αυτό το αίτημα. Ωραία λοιπόν, είναι προφανές ότι υπάρχει πλειοψηφία. μπορούμε να ψηφίσουμε για αυτή την ένσταση ονομαστικά, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Έχετε ψηφίσει όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται λοιπόν. next point. Το επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης είναι τα διάφορα, στα οποία δεν υπάρχει τίποτα. Η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει 21 και 22 Δεκεμβρίου. Ωραία λοιπόν, λίγη συνεδρίαση.